η κατάσταση των ανθρώπων με αλφισμό στην Αφρική και ιδίως στο Μαλάουι. Ονομαστική κλίση άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται το κοινό ψήφισμα λοιπόν. Κοινή κοινό ψήφισμα έξι πολιτικών ομάδων για τον Μπαχρέιν. Παράφος 2 του αρχικού κειμένου. Ψήφι υπέρ. Κατά. <clears throat> Αποχές. Εγκρίνεται. Παράγραφος 10 του αρχικού κειμένου με ονομαστική κλίση άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Ενεκρίθη. Παράγραφος 13, τροπολογία 3, ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Παράγραφος 14, το αρχικό κείμενο σε τρία τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές. Θα κάνουμε έλεγχο. Άρχεται η ψηφοφορία ελέγχου. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Ενεκρίθη. Τρίτο τμήμα. Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 4. Μονομαστική κλίση. Άρχεται η ψηφοφορία ηλεκτρονικά. Όλοι ψηφίσατε. Πέρας. Εγκρίνεται. Αιτιολογική σκέψη α, αρχικό κείμενο σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 1. Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές. Έλεγχος. Ηλεκτρονικά. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 2. Υπέρ. Κατά. Άποχες. Απορρίπτεται. Το σύνολο του ψηφίσματος όπως έχει τροπολογηθεί υπέρ. Κατά. Αποχές. Ενεκρίθη ερχόμαστε στο κοινό ψήφισμα για τη Μιανμάρ και ιδίω την κατάσταση των Ροχίνγκια. Τροπολογία 1 με ονομαστική κλίση άρχεται την ψηφοφορία. Ψήφισατε όλοι. Πέρας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 3. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 2. Ναι, θέλετε έλεγχο, βεβαίω ελέγχουμε για την 3. Αρχίτε ηλεκτρονική ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. πέρα. Εγκρίνεται. Τροπολογία 2. Υπέρ. Κατά. Έλεγχος και για τη 2. Άρχεται, είναι πολύ επικίνδυνο να εικάζει κανείς τι γίνεται. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Εγκρίθηκε. Το ψήφισμα στο σύνολό του υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Παρακαλώ. Κύριε Γκόλνης. Χωρίς μικρόφωνο ο μιλητής. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε για, το, για την ευθυδικία σας. Αναφέρομαι στο άρθρο 166 του κανονισμού που αναφέρατε προηγουμένως έναντι του συναδέλφου μου, του οποίου εγώ δεν συμμερίζομαι τις απόψεις βέβαια και δεν ανήκω στο ίδιο πολιτικό κόμμα με τον ίδιο. Αλλά θέλω να σας υπενθυμίσω κύριε Πρόεδρε ότι το άρθρο 166 σας δίνει το δικαίωμα να επιβάλλετε κυρώσει σε ένα βουλευτή ο οποίος διαταράσει σοβαρά την συνεδρία. Δηλαδή εμποδίζει τους άλλους συναδέλφου, να μιλήσουν, χειρονομεί και είσαστε υποχρεωμένοι να τον ανακαλέσετε στην τάξη. Εμένα μου έχει συμβεί αυτό μια φορά στο κοινοβούλιο κάτι τέτοιο. Αλλά το άρθρο αυτό δεν σας δίνει κανένα δικαίωμα να κολλάσετε τις δηλώσεις ενός βουλευτή ακόμα και αν έχουν χαρακτήρα εσχρό και παραβιάζουν το κοινό αίσθημα. Εγώ αν ήμουν πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου δεν θα μπορούσα να θεωρήσω, θα μπορούσα να θεωρήσω ότι κάποια πράγματα που λένε οι συναδελφοί μου είναι πραγματικά παραβιάζουν το κοινό αίσθημα ή είναι αισχρά. Αλλά υπάρχει το δικαίωμα των βουλευτών να εκφράσουν την άποψή τους και δεν έχετε το δικαίωμα τώρα να να επιβάλλετε κυρώσει σε βουλευτέ μόνο και μόνο για το περιεχόμενο των δηλώσεών του, λέει ο κύριο Γκόνη. Κύριε Γκόνης, λάβετε υπόψη στο γεγονός ότι ο κύριος Κόρβιν Μίκε είπε σε αυτήν την αίθουσα ότι είναι ουσιαστικά τα απόβλητα της Αφρικής. Αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο γίνεται αυτή η κύρωση εναντίον του και εγώ παραμένω πεπισμένος ότι είναι απόλυτα δικαιολογημένη αυτή η κύρωση. Ερχόμαστε τώρα στην έκθεση Κόβατσοφ, 71η <clears throat> Σύνοδος του, της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Πρώτη παράγραφος σε δύο τμήματα, αρχικό κείμενο. Πρώτο τμήμα υπέρ, κατά. Αποχές, εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα, υπέρ, κατά. Αποχές, εγκρίνεται. Παράγραφος ένα αρχικό κείμενο σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ, κατά. Αποχές, εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Παράγραφος 1, σημείο F, αρχικό κείμενο ονομαστική κλίση άρχεται. Ψηφίσατε όλοι, πέρας. Εγκρίθηκε. Τροπολογία 2 στην παράγραφο 1. Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται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 η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρασε. Εγκρίθηκε. Αρχικό κείμενο του σημείου W. Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Σημείο άντε με ονομαστική κλίση. Άρχεται. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. εγκρίθηκε. Το σημείο AM στην παράγραφο 1. Άρχεται η ψηφοφορία με ονομαστική κλίση. Ψηφίσατε όλοι, πέρας. Εγκρίθηκε. Το σημείο τροπολογία 8. Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Λοιπόν, σηκώντε τα χέρια όμως σας παρακαλώ. Τροπολογία 8, ηλεκτρονική επαλήθευση. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Εγκρίθηκε. Τροπολογία 4. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Το αρχικό κείμενο στο ΑΠ. Υπέρ. Κατά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 το αρχικό κείμενο στο σημείο AV σε τρία τμήματα. Πρώτο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τμήμα 2. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τρίτο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. AW στο αρχικό κείμενο σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτό. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 6 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 7 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Το ψήφισμα ως σύνολο με ονομαστική κλίση άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρασε προφορία. Εγκρίνεται η αχθιστικό. Κόμετσεφ. Ερχόμαστε στην έκθεση της κυρίας Στίβενς για την εφαρμογή της σύμβασης του ΟΗΕ για τα δικαιώματα των ανθρώπων με αναπηρίες. Παράγραφος 1 σε δύο τμήματα πρώτο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Παράγραφος 15. Ε, Αρχικό κείμενο σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Παράγραφος 16. Αρχικό κείμενο σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχέ εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχέ Εγκρίνεται. Παράγραφος 25. Αρχικό κείμενο σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχέ. Εγκρίνεται. Παράγραφος 28. Αρχικό κείμενο υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Παράγραφος 31. Σε δύο τμήματα. Το αρχικό κείμενο υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές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 αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Ε, ηλεκτρονικός έργος για την 110 δεύτερο τμήμα. Ψηφίσατε όλοι. Ψηφίσατε όλοι. Πέρασε. Απερίφθη. Παράγραφος 116. Σε δύο τμήματα με ονομαστική κλίση και τα δύο. Πρώτο τμήμα άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα πάλι ονομαστική κλίση άρχεται. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Απορρίπτεται. 118 Αρχικό κείμενο. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 127 σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά. Απόχε. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές. Ελέγχουμε. 127 δεύτερο τμήμα. Ηλεκτρονικά. Άρχεται η ψηφοφορία. Σφίσατε όλοι. Πέρας. Με μία ψηφοδιαφορά απορρίπτεται. 147 αρχικό κείμενο υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 149 σε δύο τμήματα πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχέ εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 165 σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται έλεγχος 165 τμήμα 2 <clears throat> άρχεται ψηφίσατε όλοι πέρας εγκρίνεται Αιτιολογική σκέψη Z σε δύο τμήματα με ονομαστική κλίση και τα δύο. Πρώτο τμήμα. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα. Με ονομαστική κλίση άρχεται. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. εγκρίνεται. Αιτιολογική σκέψη ΑΑ. Αρχικό κείμενο, ονομαστική κλίση δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα, άρχεται η ψηφοφορία. Σφίσατε όλοι πέρας. Εγκρίθηκε. Δεύτερο τμήμα, πάλι ονομαστική κλίση. Άρχεται. Σφίσατε όλοι. Πέρας. Απορρίπτεται. Ωραία. Τελική ψηφοφορία, το σύνολο όπως έχει τροποποιηθεί, ονομαστικά. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Εγκρίνεται. αντίληψη βάσει του άρθρου 106 για επιτρεπόμενες, επιτρεπόμενες ισχυρισμοί στα τρόφιμα. Παράγραφος 4 μονομαστική κλίση. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 20 Κατά. Αποχές. Εγκρίνονται. 21. Αρχική, αρχική περκόκιμο υπέρ κατά <clears throat> αποχές. Απορρίπτεται. Αιτιολογική σκέψη α. Αρχικό κείμενο. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Να το ελέγξουμε. Άρχεται η ηλεκτρονική ψηφοφορία. Ψήφισαν όλοι. Πέρασε. Εγκρίνεται. Τροπολογία 5. Υπέρ κατά αποχές. Ελέγχουμε την 5. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψήφισατε όλοι πέρας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 6. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Αν δεν σηκώσετε τα χέρια δεν μπορώ να σας δω. Θα αναγκαστούμε να ελέγξουμε. Μάλιστα. Αρχίζουμε. Ψηφίσατε όλοι. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Εγκρίνεται. Αιτιολογική σκέψη B. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Ελέγχουμε. Ηλεκτρονική ψηφοφορία για την αιτιολογική σκέψη B. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 1. <clears throat> Ονομαστική κλίση. Αρχίζει η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Απορρίβεται. Αρχικό κείμενο στην αιτιολογική σκέψη τσε. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. <clears throat> Τροπολογία 2. Υπέρ. Κατά. <clears throat> αποχές εγκρίνεται καλά να ελέγξουμε όπως θέλετε αφού αγαπάτε αρχίζει η ηλεκτρονική ψηφοφορία ψηφίσατε όλοι πέρας <clears throat> Εγκρίντη. τροπολογία 11 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 12 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 13 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 22 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται τροπολογία 7 <clears throat> υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται τροπολογία 8 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 9 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 10 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται